Τροπολογία 5. Το πρώτο τμήμα το ψηφίσαμε. Τώρα θα ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Το δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας 5. Κατά. Αποχές δεκτό. 23. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα συνεχίσουμε ε, σύντομα την ψηφοφορία. Να σας ξαναπώ ότι δεν αναφέρω τα δύο πρώτα ψηφία, δηλαδή το 6 και το 0, το 60. Θα λέω τα δύο τελευταία ψηφία. Οπότε τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 6. Η κυρία Γκαρσία Περέζ. Θέλουμε να γίνει έλεγχος ηλεκτρονικός στην 24. Μάλιστα. Να γίνει. Τροπολογία 24. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Επιβεβαιώνω ότι οι συνάδελφοι ΕΛΚ δεν ψήφισαν τις προηγούμενες τροπολογίες, δεν πρόλαβαν. Είμαστε ακόμα στην αρχή της διαδικασίας. Έχετε την καλοκυσίνη να ξαναρχίσετε από την αρχή γιατί υπήρξε μια μικρή παρανόηση. Το ξέρω, Πρόεδρε. Αλλά δεν ψηφίσαμε. Λυπάμαι. Δεν μπορούμε να ξανά κάνουμε παλιές, άλλες τις ψηφοφορίες που τις είχαμε κάνει. Ξεκινάμε με την τροπολογία 24, τώρα, άρχεται η ψηφοφορία. Το ΕΛΚ έχει δύο, δύο παραπάνω ψήφους.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 I'm so sorry, we can't vote. δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Διότι... Voting. And... Η ομάδα Freedom με Democracy έχει δύο επιπλέον μέλη. Δεν μπορούμε. Μόνο ε, επιτροπή, μέλη της Επιτροπής Γενικών ψηφίζουν για τον προπολογισμό. Freedom με Democracy έχουν δύο επιπλέον. Πρέπει να βγουν αυτά. We try to do a new start and I'm sorry. Αρχίζουμε και λυπάμαι. Θα πρέπει να ξαναψηφίσουμε την τροπολογία 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι τα ίδια. Έχουμε... Υπάρχει μια... ένας επιπλέον ψήφος. Δύο μάλλον. Πώς να σας το πω. Δύο από την ομάδα Freedom Democracy, δύο μέλη θα πρέπει να φύγουν. Μόνο η Επιτροπή Γυναικών ψηφίζει. Πώς να το κάνουμε. So that we Ε, και έτσι καθυστερούμε. Λυπάμαι για αυτό το πρόβλημα, αλλά τι να σας πω. Ρόμεν Ρόιτεν. E Για να ελέγξετε κύριε Πρόεδρο ποιος είναι παρόν από αυτή την ομάδα. Και να, άμα είναι να, να, να μάθουμε ποιο χρειάζεται να βγάλει την κάρτα του και άμα να συνεχίσουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, θα το πράξουμε τώρα. Θα το δούμε.

Για να σηκώσουν τα χέρια τους, τα μέλη. Από την Επιτροπή, από την ομάδα Ελευθερία και, Δημοκρατία. Α, τέλος πάντων, ξεκινάμε. Άρχεται η ε, ψηφοφορία 24. still two members. Πάλι τα ίδια. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. τώρα θα και ψηφίζομαι ηλεκτρονικά και θα βγάλουμε τα δυο ονόματα από την ομάδα EFD. Λοιπόν, ξαναψηφίστε την τροπολογία 24, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Είναι ξεκάθαρο ότι απορρίπτεται. Προχωρούμε. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26. Φιγκερέδο. Υπέρ. Πάμε πίσω και ελέγχουμε την 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 6. Της Γκαρσία Περέζ. Α, δεν λειτουργεί το μηχάνημα το ένα. Ξαναρχίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 6. Πέρασε. Απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έλεγχος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Περσέβει μία ψήφος του ΕΛΚ. Εντάξει, βρέθηκε. Πέρας. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία, τροπολογία 8. Πέρας. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 12. Α, να με το κείμενο της 11. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτό και το κείμενο. 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Πάμε στη 13. Γκαρσία Περέζ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ καταπίπτει οπότε πάμε στην 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή Α, ελέγχουμε την 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Περσέβει μια ψήφος του ΕΛΚ. Τώρα είναι εντάξει. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται 28. Πάμε στην 29. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Όχι, έλεγχος. Ελέγχουμε την 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Περσεύει μια σοσιαλιστική ψήφος, παρακαλώ. Κοιτάξτε το, τώρα είναι εντάξει. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 30 με προφορική τροπολογία. Δέχεστε την προφορική τροπολογία. Ναι. Ψηφίζουμε την 30 λοιπόν με την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή αυτό ε, ήταν, τελειώσαμε. Συγγνώμη για τα προβλήματα στην ψηφοφορία. Υπήρξε κάποια σύγχυση. Ευχαριστώ. Επομένως, να ξεκινήσουμε με την κοινή μας συνεδρίαση, με την, ε, με την ε, Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Θα ήθελα να χαιρετήσω ε, όλους τους συναδέλφους και εκ μέρους ε, το, εδώ της γραμματείας όλους συναδέλφους, συναδέλφισες και διερμηνείς να τους χαιρετήσω, να τους καλωσορίσω σε αυτήν εδώ τη συνεδρίαση. Καταρχήν να εγκρίνουμε την ε, ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν προτάσεις ε, για αλλαγές, οπότε θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Ε, τα, τα πρακτικά από τις 20 Δευτέρα Ιουνίου τα έχετε στη διάθεσή σας. Αν δεν υπάρχουν σχόλια θα θεωρηθούν ότι εγκρίνονται έχουμε να κάνουμε με την εμπορία ε, παράνομη διακίνηση ε, ε, ανθρώπων. Υπάρχει η οδηγία της Επιτροπής για αυτό το θέμα. Ένα θέμα στο οποίο κυρίως ή μάλλον ένα μέρος αυτού του προβλήματος αφορά παιδιά και γυναίκες αυτό το θέμα βρίσκεται στην αρμόδιότητα τόσο της δικής μας Επιτροπής αλλά και της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, αποφασίσαμε να κάνουμε μια κοινή συνεδρίαση σύμφωνα με το κανονισμό του άρθρο 51. Είχαμε ένα κοινό σεμινάριο όπου είχαν, οι συνάδελφοι και από τις δύο επιτροπές είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν αυτό το θέμα. 13 Ιουλίου είχαμε μια παρουσίαση από τους ε, αρμόδιους Σήμερα έχουμε μια ενδεικτική θα λέγαμε ψηφοφορία για να έχουμε μια εντολή στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν με το Συμβούλιο. Εγώ χαίρομαι που μπορούμε να πούμε είχαμε μια πολύ αγασή συνεργασία ανάμεσα στις δύο εισηγητές των δύο επιτροπών και εν γέννη με την Επιτροπή την, των Δημοσίων Ελευθεριών με τη γραμματεία τους πραγματικά μια πολύ σωστή συνεργασία. Και πριν να περάσουμε σε αυτήν θα, θα λέγαμε την ενδεικτική, την κατευθυντήρια ψηφοφορία θα ήθελα να δώσουμε το λόγο στους δύο εισηγητές, συγγήτριες ε, και θα αρχίσουμε με την κυρία Μπάουερ από την Επιτροπή Γυναικών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εξηγήσω μια συνήθιστη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε εδώ, γιατί συνήθως γινόταν συζήτηση για τις τροπολογίες. Όμως, η κατάσταση είναι ως εξής. Στις θερικινές διακοπές δεχτήκαμε πάνω από 200 τροπολογίες και ήταν αδύνατον να συζητήσουμε με όλους τους εμπλεκομένους όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ζητώ συγγνώμη και εγώ και η συνάδελφος γι' αυτό. Δεχτείτε λοιπόν αυτήν την έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ για την εξαιρετικά καλή συνεργασία. Βλέπετε τα αποτελέσματα. Συμφωνήσαμε στο 90 σχεδόν της 100 επί του καταλόγου των ψηφοφοριών με την σοσιαλίστρια συνάδελφο από τη Λίμπε αλλά χωρίσαμε ε, την ψηφοφορία ανάλογα με τις πολιτικές ομάδες και τις επιτροπές και καλώ τους συναδέλφους από το ΕΛΚ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να ακολουθήσουν τον κατάλογο ψηφοφοριών της Επιτροπής ΦΑΜ. Ευτυχώς ε, είμαι υπεύθυνη ισχυώδης εισηγήτρια στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και για το ΕΛΚ. Για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ επίσης για την εξαιρετικά καλή συνεργασία και με τις δύο γραμματείες και με τις δύο εκπροσώπους και τις υπεύθυνε. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία μας και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χέντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύντομα να πω ότι 100% υποστηρίζω αυτά που είπε η κυρία Μπάουερ και τα ευχαριστώ σε όλους όσους συνεργαστήκανε μαζί μας. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Είναι ένας μεγάλος αυτός δρόμος, αλλά αν συνεχίσει το ίδιο καλά νομίζω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή ε, νομοθεσία. Ε, θα επανέλθω κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Ανακαλύψαμε ότι η συμβαστική ε, τροπολογία 21 της συναδέλφου σας Μπουσκούτ δεν συμπεριλαμβάνει όλη την ε, τροπολογία 95 ε, και εκεί θα θέλαμε ε, να κάνουμε μια χωριστή ε, ψηφοφορία. Αλλά αυτό θα το δούμε όταν φτάσουμε στην συμβαστική τροπολογία 21. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε την κυρία Χέντ. Η κυρία Αργεντίνη ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στο Συμβασμό 21 η τροπολογία μας υπαριθμών 98 για την τήρηση των αρχείων δεν περιλαμβάνεται στο Συμβιβασμό 21. Θα υποβάλω προφορική τροπολογία διαφορετικά. Θέλω να ψηφιστεί η δική μας, η 98. Θα ψηφίσουμε επί της τροπολογίας αυτής του, της 98. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία και να επενθυμίσω ότι είναι, ε, θα λέγαμε, ενδεικτική ε, αυτή η ψηφοφορία και χαίρομαι που μοιράζουμε την Προεδρία σήμερα με τον κύριο Λόμπερς Αγιλάτο που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Τον ευχαριστώ πριν να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Πιστεύω ότι όλοι είναι έτοιμοι και μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Αρχίζουμε με την 116 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκατόν δέκα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά χες εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 122. Αρχίζει η ψηφοφορία. with the technicians. We must check with the... Δεν ξέρω που έγκυται το πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. I'm so sorry, but it's some problem. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρα σας παρακαλώ διανατάσεως ψηφίζουμε την 122. Ποιοι είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Against. Κατά. Εγκρίνεται. Έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Γι' αυτό έγινε καταμέτρηση και υπάρχει πλειοψηφία. Έξι επιπλέον υπέρ, άρα εγκρίνεται. Ελπίζω το θέμα να επιληθεί. Τώρα φτάνουμε στο συμβασμό 2, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ όχι καταπίπτει. 130 υπέρ παρακαλώ 130 ψηφίζουμε τελικά υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Η κυρία Παρβάνοβα. Έχουμε μία προφορική και τρεις οριζόντιες που έχουν ενταχθεί στο τέλος, αλλά θα πρέπει να ψηφιστούν εδώ. Μπορούμε καταρχήν να ψηφίσουμε την προφορική που βρίσκεται στο τέλος του καταλόγου, γιατί αφορά την 121, 175, 160 και, την, και το συμβασμό 6. Αυτές οι τρεις οριζόντιες βρίσκονται στο τέλος, αλλά φορούν την παρούσα. Ναι, κυρία Παρβάνοβα, μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα και θα βρείτε στη σελίδα 21 νομίζω τις τροπολογίες αυτές. Στην τελευταία σελίδα έχετε τις τρεις οριζόντιες προφορικές. Βρήκατε, τις βρήκατε, τις βρήκατε, τις τρεις προφορικές από τους φιλελεύθερους. Η πρώτη προφορική υπέρ, παρακαλώ, υπέρ της πρώτης προφορικής κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη προφορική από τους φιλελεύθερους υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και έχουμε και μία προφορική από τους πράσινους. Μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα, επανερχόμαστε στην 131. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ναι, κυρία Μπάουερ, ψηφίζουμε τις 21, την 21, 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την 132. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, ζητήστε το λόγο γιατί ακούω παρατηρήσεις αλλά εκτός μικροφώνου. Εντάξει. Κυρία Παρβάνοβα, ζητήσαμε, ελέξουμε ηλεκτρονικά την 131. Ωραία. 131, ας προσπαθήσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 131. Απορρίπτεται. 15 υπέρ, 34 κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 132 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 23 αποσύρεται, άρα ψηφίζουμε την 133 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια έχουν την τροπολογία 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132, 142 με συγχωρείτε. Α, με συγχωρείτε λέει η πρόεδρος για τρίτη φορά έκανα λάθος. 141 141 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, θέλετε να ελέγξουμε, εντάξει. Ελέγχουμε την 143, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 31 υπέρ. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 151 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές να ας ελέγξουμε 153 ελέγχουμε ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. 154 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβασμού 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 163 αρχίζει η ψηφοφορία. πέρα. εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. 21 κατά. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ. Θα ήθελα να προβάλλω μία προφορική στην 165, άρθρο 10, παράγραφος 5. Θα ήθελα να προσθέσουμε μετά το κείμενο τα κράτη-μέλη θα δράσουν σύμφωνα με την ε, οδηγία του Συμβουλίου 2004-81, δηλαδή ως προς την άδεια παραμονής, χορήγηση άδειας παραμονής. Υπάρχουν αντιρρήσεις με την ε, προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Κυρία Μπάουερ, καλύπτεται από την 162, η οποία και εγκρίθηκε. Καλύπτεται αυτό το θέμα. Άρα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, αλλά είχαμε μία επεξήγηση από την κυρία Μπάουερ. Άρα ψηφίζουμε την 165. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 166. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 167. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. ψηφίσουμε την 168 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 160, 170 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. 176 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 27 υπέρ, 21 κατά. 177 υπέρ, κατά αποχές ας ελέγξουμε 177 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 27 υπέρ 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ 80 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα έχουμε την τροπολογία συμβιβασμού υπαριθμών 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε, ωραία, ελέγχουμε την 192, αρχίζει η ψηφοφορία. Για την 192. Πέρας εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ. 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στη 200 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 συμβιβασμού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Θέλετε να ελέγξουμε. Εντάξει, ελέγχουμε γιατί τη 204. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 21 ψήφι κατά 24 υπέρ, 24 κατά, 205 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 45. Το πρώτο τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται. 207 τώρα ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Α, 210 το πρώτο τμήμα υπέρ Θέλετε να ελέγξουμε την 209, εντάξει. 209 της κυρίας Head. 209 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται με 32 ψήφους υπέρ. 210. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε το, 210 το δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 218 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 221 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 223 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές ε, ε απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 συμβιβασμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ Θέλετε να ελέγξουμε την 61. Ελέγχουμε για την 61. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. Η 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα. 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε. 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Συμβιβαστική 16. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τώρα η τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές δεκτή 90 υπέρ κατά αποχές δεκτή 91 υπέρ κατά αποχές δεκτή τώρα συμβιβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή η 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική 21. Η κυρία Χέντε έχει το λόγο, παρακαλώ. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που έλεγα πριν για την 95 τροπολογία που δεν καλύφθηκε. Θέλουμε χωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία 95 λοιπόν. Κυρία Χέντ, για εξηγήστε μας συγκεκριμένα. Γιατί θέλετε χωρίς τη ψηφοφορία. Παρακαλώ, κυρία Χέντε. Είναι το πρώτο τμήμα, όχι το, δεύτερο τμήμα, για τη δέουσα επιμέλεια στον εντοπισμό και την εξάλληψη της ανάμειξης ή συνενοχής του δημόσιου τομέα στην εμπορία ανθρώπων. Ωραία. Οπότε κατατοπιστήκατε για την 95 που θα ψηφιστεί χωριστά. Ψηφίζομαι. Τροπολογία 95. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα. Τώρα θα ψηφίσουμε τη συμβαστική 21. Μισό λεπτό. Ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εγώ ζήτησα για την 98 χωριστή ψηφοφορία γιατί δεν νομίζουμε ότι καλύπτεται από τη συμβιβαστική 21 και χωριστά εκεί που λέει ε, με, σε πνεύμα πλήρου σεβασμού του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Είναι το δικαίωμα του προσώπου ε, του οποίου δεδομένα συλλέγονται. Πρώτα θα ψηφίσουμε λοιπόν όλη τη συμβαστική 21 και μετά θα ψηφίσουμε την 98. Μα γιατί, αφού την 95 την, τώρα την ψηφίσατε από πριν, γιατί και αυτοί μερικοί θεωρούσαν ότι καλύπτεται από τη συμβιβαστική 21. Α, παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Εντάξει, εντάξει. Ψηφίζομαι την συμβιβαστική 21 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα ψηφίζομαι την 98 τροπολογία και ακούσατε την εξήγηση. Ψήφι υπέρ της 98 κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και πάμε στην 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 100 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 101 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 15. Α, έλεγχος Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την τροπολογία 103. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται, συγγνώμη, είπε, ότι εγκρίνεται η πρόεδρος. Όχι, όχι. Ε, απορρίπτεται. 21 ψήφοι υπέρ, 25 κατά απορρίπτεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 106 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 108 Α, θα ελέγξουμε την 107 ηλεκτρονικά, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 113 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 115 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Θέλετε έλεγχο. Τη 115 ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Δεκτή. Με 26 ψήφους υπέρ και 19 κατά. Και τώρα Τελική ψηφοφορία. Πρόταση της Κομισιόν ως ετροποποιήθη. Τίθεται σε ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 42 ψήφι υπέρ, μία ψήφος κατά, πέντε αποχές. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στις εισηγήτριες και ευχαριστούμε και όλες και όλους για την υπομονή κατά την ψηφοφορία που ήταν λίγο προβληματική στην αρχή. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή συνεργασία όλους και όλες.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 Καθίστε παρακαλώ. Πρέπει να συνεχίσουμε. Καθίστε, συνάδελφοι, και αν θέλετε να συνομιλήσετε με κάποιον, να το κάνετε εκτός εθούσης. Τώρα συνεχίζουμε την κοινή μας συνεδρίαση ε, και θα δούμε ένα άλλο θέμα, την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Σύμφωνα με τον κανονισμό άρθρο 51 έχουμε ένα κοινό έργο, οι δύο επιτροπές και αυτό και αυτό το μέλος τη συνεδρίαση θα γίνει με προεδρία από κοινού. Ε, θα έχουμε την κυρία Λότης Αγγιλάρ μαζί μας. Συγγνώμη, τον κύριο Λότης Αγγιλάρ. Είναι μια πρωτοβουλία για να μπορέσουμε να πετύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την εντολή προστασίας. Ο στόχος με αυτήν εδώ την πρωτοβουλία είναι να προστατεύσουμε θύματα ακόμα ακόμα κι αν ένα θύμα ε, βρίσκεται σε μια άλλη χώρα από τη χώρα από την οποία κατάγεται. Εμείς Είχαμε κοινέ συζητήσεις ε, παλαιότερα στις δύο επιτροπές. Υπάρχει η 12η Ιουλίου που ήταν ε, η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. Έχουμε 141 τροπολογίες και ο στόχος της σημερινής συνεδρίασης είναι να συζητήσουμε αυτές εδώ τις τροπολογίες. Εγώ θα ήθελα να δώσω το λόγο και στις δύο εισηγήτριες. Οι Σιμινές είναι από Επιτροπή Γυναικών και η κυρία Ρομέρο από την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Πρώτα θα δώσω το λόγο στην κυρία Χιμενές. Παρακαλώ. Ξεκινά. Buenos días. Καλημέρα σας. Έγινε λόγος για ένα μεγάλο αριθμό τροπολογιών. Δεν θα τις αναφέρω. Κάτι το οποίο καταδεικνύει ότι κανείς δεν είναι αδιάφορος και η εργασία μας στις χώρες μας υπέρ των θυμάτων βίας ε, την χάνει μια κοινή προσέγγισης από το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένα πολύ καλό μέσο έτσι ώστε τα θύματα βίας να αισθανθούν ότι προστατεύονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας πω, μελετώντας τις τροπολογίες, ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ θετικό, αλλά θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι παρά τις τροπολογίες ε, που λάβαμε που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ε, Ευρωεντάλματος θα πρέπει να μας απασχολήσουν έτσι ώστε τα θύματα βίας να την χάνουν τις προστασίες που χρήζουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους διότι εμπλούτησαν αυτή την έκθεση με τις τροπολογίες και σας είπα πολλές φορές ότι ο δρόμος μας δεν ήταν εύκολος γιατί υπάρχουν διαφορετικές ε, νομοθεσίες στα κράτη-μέλη και αυτό είναι το μεγάλο πρόσχημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να μετατραπεί το ευρωένταλμα σε πραγματικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας και ο νόμος θα πρέπει να γνωρίζει τις ελευθερίες κάθε κράτους. Θα ήθελα να πω ότι κάθε κράτος αναγνωρίζει πότε ένα θύμα πρέπει να τύχει προστασίας. Γι' αυτό θα βρούμε και λύσεις έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά των τροπολογιών. Θα το κάνουμε διότι το χρωστάμε στα θύματα. Θα πρέπει να πηλήσουμε τις διαφορές μας, να έχουμε ένα μέσο το οποίο να είναι σαφές και ε, να μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα. Πρόκειται για μία φιλόδοξη εντολή και είμαι πολύ ευχαριστημένη με τις τροπολογίες. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας, του δουλεμπορίου και της, του μαδικού εγκλήματος. Παιδιά τα οποία γνωρίζουν βία και γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε και για προγράμματα πρόληψης και πληροφορίας στα κράτη-μέλη και άλλες ε, βελτιώσεις που δεν θα ήθελα να ε, αναφέρω διότι δεν έχουμε ε, χρόνο. Θα το συζητήσω διμερός με όποιον το επιθυμεί. Ελπίζω σε, με αυτή τη διαπραγμάτευση να βελτιώσουμε ορισμένες τροπολογίες που δεν είναι αναγκαίες και αναφέρονται στη νομική βάση. Επίσης ε, θα πρέπει να αιτιολογήσουμε την απόρριψη, την τυχόν απόρριψη εφαρμογής αυτής της ε, ευρωεντολής. Γιατί ό,τι θεωρείται έγκλημα σε μία χώρα, ίσως να μην θεωρείται σε μία άλλη. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, διότι το οφείλουμε στα θύματα βίας. Νομίζω λοιπόν ότι στις 29 θα ψηφίσουμε για να μην ξεχνάμε το, το βασικό μας μέλημα που είναι η ασφάλεια των πολιτών. Θα είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή την, για αυτή την έκθεση γιατί παρά τις επικρίσεις εμπλουτίσαμε το περιεχόμενο και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι αν εγκριθεί ότι επιλύσαμε πολλές διαφορές και διευκολύναμε τη ζωή των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Χιμινές και, θα αμέσως θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρομέρο. Παρακαλώ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας και διότι έτσι καταφέραμε να βελτιώσουμε το κείμενο και θα ήθελα να πω ότι το άρθρο 1 είναι επίμαχο, δηλαδή το, το πεδίο εφαρμογής. Πιστεύω ότι αυτή η ευρωεντολή θα πρέπει να ψηφιστεί από όλους διότι ο πυρήνας του ζητήματος είναι το εξής. Υπάρχουν χώρες που χρησιμοποιούν μία νομοθεσία προληπτικής φύσης, δηλαδή μέτρα αστυνόμευσης και διοικητικά, μέτρα που κινούνται πολύ πιο γρήγορα από τις δικαστικές αποφάσεις που αργούν ιδιαίτερα θα πρέπει να προσβλέπουμε προς αυτές τις χώρες που ακολουθούν αυτή την ε, γρήγορη διαδικασία για να προλάβουν την δολοφονία γυναικών. Αυτά τα αστυνομικά ή διοικητικά μέτρα όμως προτρέχουν των δικαστικών αποφάσεων και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να φτάσουμε σε μία συμφωνία. Διότι εάν αναμένουμε μία δικαστική απόφαση, τότε το έγκλημα ίσως έχει ήδη λάβει χώρα. Άρα δεν δρούμε εγκαίρως. Όποια και να είναι η νομοθεσία προληπτικής φύσης, γιατί ξέρουμε ότι η δικαιοσύνη αργεί ιδιαίτερα, όποιο προληπτικό πλαίσιο λοιπόν και να εφαρμοστεί, θα πρέπει να εγγυηθούμε την προστασία του θύματος. Γι' αυτό το πεδίο εφαρμογής δεν μπορεί να λάβει υπόψη τα διαφορετικά παραδοσιακά συστήματα δικαιοδοσίας εάν δεν λάβουμε υπόψη την προστασία του θύματος. Γνωρίζουμε ότι, θα, ότι η Επιτροπή αντιτίθεται. Άρα στο άρθρο 3 της συνθήκης θα πρέπει να προβάλλουμε τις αιτιολογικές σκέψεις όπως θέλει και η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Διότι η ελευθερία κυκλοφορίας θα πρέπει να ισχύει και για εκείνους που αποτελούν αντικείμενο βίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επόμενη συμφωνία του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης. Γι' αυτό ό,τι αποφασίσει το ε, Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να αποστείλουμε ένα ε, μήνυμα υπέρ της προστασίας των θυμάτων όπου και να βρίσκονται. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε τα 27 κράτη-μέλη προ των ευθυνών τους. Υπάρχουν πολλά που προβάλλονται από τις ε, τροπολογίες, πολλά επιμέρους ζητήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ε, διεθνικές, διακρατικές ε, τροπολογίες, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια συνολική συμφωνία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ρομέρα. στην, στον κατάλογο εμιλητών έχει το λόγο. Ja, vielen äh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εισηγήτριες καταρχήν που έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά. Γιατί εδώ πραγματικά δηλαδή έγινε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Αφενός υπάρχουν διάφορα δικαιικά συστήματα στα κράτη-μέλη. Αφετέρου Μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε να δημιουργήσουμε ή δυνατόν ένα πλαίσιο για την παροχή βοήθεια στα θύματα. Στις επικείμενες διαπραγματεύσεις πρέπει οπωσδήποτε να παλέψουμε ώστε η νομοθετική πρόταση για συνεκτικό μέσον ε, να γίνει υπέρ των θυμάτων και γι' αυτό πρέπει να πείσουμε πολύ κόσμο ακόμα. Ο συνάδελφος Τριανταφυλλίδης και εγώ επικεντρωθήκαμε άλλη μια φορά στα θέματα που προκύπτουν από τις τροπολογίες ως σκιώδης από την ομάδα μας για τις Επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΦΑΜ. Είναι σημαντικό ότι θα πρέπει να είναι εγγυημένη η προστασία για όλα τα θύματα. Αυτό προσπαθούν και οι συγγήτριες, αυτό, σε αυτό αποσκοπούν και οι τροπολογίες είναι σημαντικό η φυλετική διάσταση να είναι οριζόντια και εδώ πολλά μπορούμε να βελτιώσουμε. Επίσης σημαντικό είναι, το θέμα της προστασίας των ανηλίκων και θέλουμε, και αυτό είναι επίμαχο θέμα, ε, θέλουμε να μην προκύψουν πρόσθετες δαπάνες για τα θύματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ. Παραδιάσεις κατά των διατάξεων προστασίας και εδώ υπάρχει κάποια αταξία και θα πρέπει να τα συζητήσουμε και να δούμε πώς θα, θα αντιμετωπίσουμε τις παραβιάσεις και τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί υπάρχουν διάφορες προτάσεις μέσα από τις τροπολογίες. Πολύ σημαντικό είναι για μας και υπάρχουν εδώ σημαντικές βελτιώσεις μέσα από τις τροπολογίες και ε, συμφωνούν οι συγκήτριες ότι οι δράστες δεν πρέπει να έχουν επαφή, ε, δυνατότητα προσέγγισης των θυμάτων. Ε, αυτό δεν πρέπει να γίνει με κανένα τρόπο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να προσεγγίζουν τα προστατευόμενα πρόσωπα. Πολύ σημαντικό είναι επίσης και υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις εδώ το θέμα των συλλογών πληροφοριών, δεδομένων και το θέμα της προστασίας τους. Δεν θέλουμε δηλαδή καρτέλα θυμάτων, ε, ε, κατάστοιχα θυμάτων αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται να υπάρχουν δεδομένα. Τέλος, η προθεσμία για την εκτέλεση άμεσα, 15-20 μέρες, άμεσα, άμεσα σημαίνει άμεσα. Εγώ συμφωνώ, ε, αλλά θα το δούμε και κατά τις ψηφοφορίε και κατά τις συζητήσεις. Και άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ από την ομάδα μας προς τους εισηγητές. Ευχαριστούμε την κυρία Ένστ. Στον κύριο Λακολίνο τώρα ο λόγος. Στο κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ τις δύο εισηγήτριες για το έργο που κάνανε. Πραγματικά κάνανε μια προσέγγιση πολύ μετρημένη σε ένα δύσκολο και περίπλοκο θέμα. Μην ξεχνάμε, στην τελευταία συνεδρίαση, η ε, μην ξεχνάμε, ε, ξεχνάμε δηλαδή που είχαμε συζητήσει για το ότι η, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ήταν με την Ισπανία και την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ προσπάθησε να κάνει σοβαρή ε, δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. αυτή η απόφαση για προστασία σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο ε, είναι ένα θέμα που μιλάμε, μιλάνε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, χωρίς καθυστέρηση. Ε, αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξουν εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις. Ούτως ώστε να προχωρήσουμε ε, σε μια απόφαση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε μια καθυστέρηση μπορεί να είναι επικίνδυνη λένε ότι ένα αρχείο είναι απαραίτητο, ένα μητρό. Όχι, δεν συμφωνώ. Μπορεί να είναι χρήσιμο, ενδεικτικά έστω, για να δίνει πληροφορίες στις αρχές. Για μένα είναι απαραίτητο. Και τα μέτρα προστασίας του ατόμου θα πρέπει να γίνονται στα μέτρα της προστασίας της οικογενείας του θύματος. Θα πρέπει να προβλεφθεί και αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γιανακουδάκη είναι η επόμενη ομιλήτρια. Um, Ευχαριστώ. Καταρχήν ο Σκιώδης πολύ γρήγορα για την Επιτροπή ΦΑΜ. Συμμερίζομαι τα συναισθήματα της εισηγήτριας από την ομάδα μας. Ελπίζω κάποια μέρα αυτή η εντολή προστασίας να υπάρξει. Είναι σημαντικό να είναι οι βασικές γραμμές τις σωστές. Αυτό είναι η βασική μου ανησυχία. Εκπροσωπώ τον Τίμωθη Κάρτο που είναι ο σκιώδης για τη Λίμπε και ο οποίος έπρεπε να πάει στη διάσκεψη των Προέδρων μ' άφησε την ομιλία του. Οπότε παραθέτω διαβάζοντας, είναι ε, δικηγόρος και το βλέπει από τεχνικής άποψης. Ο Τίμωθη λέει λοιπόν, πιστεύουμε ότι τα θύματα οικιακής βίας και άλλων ε, αξιόπινων πράξεων θα πρέπει με εμπιστοσύνη να διακινούνται στην Ευρώπη, γνωρίζοντας ότι θα έχουν παντού προστασία. Θέλουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους να συνεργαστούμε για να το καταφέρουμε αυτό. Καταρχήν χαιρετίζομαι τους στόχους της Ευρωπαϊκής Εντολής Προστασίας. Υπάρχουν όμως κρεμή θέματα που αφορούν νομική βάση, πεδίο εφαρμογής του μέσου, που απειλούν να υπονομεύσουν κατά την ε, έγκρισή του το μέσο. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά πάνω στο κείμενο για να ασχοληθεί με τα προβλήματα αυτά. Θα ήθελα να παρουσιάσω τα βασικά μας προβλήματα εν συντομία. Πρώτον, Πιστεύουμε ότι η έκθεση αυτή, ως έχει αυτή τη στιγμή, ξεπερνά το πεδίο εφαρμογής μιας ε, ε, νομικής ε, βάσης για ποινικά θέματα. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δεύτερον, οι τροπολογίες 89 με 92 προτείνουν να χρησιμοποιηθεί η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη δεν έχει νομοθετική νομική βάση. Αυτό είναι ανησυχητικό δεν μπορούμε το, να έχουμε νοσιακό δίκαιο χρησιμοποιώντας μέσων που στερείται νομικής βάσης. Τρίτον, οι 215, 216, 217 και 218 θέτουν το ζήτημα των χρονικών περιθωρίων ενώ τα χρονικά όρια και περιθώρια και προθεσμίες είναι σημαντικά, δεν μπορούμε να ζητήσουμε να θεσμοθετηθούν οι προθεσμίες αυτές. Τέλος, οι 105, 106 και 228 αφορούν στο γεγονός ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλονται δαπάνες στα προστατευόμενα πρόσωπα. Δεν, δεν συμφωνούμε, πιστεύουμε, ότι θα πρέπει να αφήνεται αυτό στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, να καθορίζουν τυχόν δαπάνες. Αυτά λέει ο Τίμωθη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Γιάννα Κουδάκη. Η κυρία Κώστα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια οι συγγήτριες σε ένα θέμα το οποίο θα λέγαμε ότι είναι ναρκαπέδιο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι καιρός οι χώρες μέλη να ε, περάσουν αυτή την πρωτοβουλία ε, στο Συμβούλιο και εδώ πέρα έχουμε ένα μεγάλο αίτημα ε, και δι των γυναικών στις χώρες μας. Ξέρουμε ότι όλες οι χώρες Ευρώπης ή σχεδόν είναι υπέρ μιας νομοθεσίας όλο και πιο προχωρημένες για να προστατεύσουν τα θύματα και να ε, προλάβουν όλους τους τύπους βίας. Ε, ε, το βλέπει κανείς η νομοθεσία το θέμα της προστασίας σε σχέση με τη βία, αλλά υπάρχει μια ανισότητα στη χώρα μου. Φερπίνη. Υπάρχει η παρέμβαση, ε, η δυνατότητα να προστατεύσει κανείς τα, το θύμα. Ε, φυσικά από χώρα σε χώρα υπάρχουν αλλαγές, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι η καλύτερη λύση είναι να δουλέψουμε συντονισμένα και να προχωρήσουμε ε, σε επίπεδο νομικό έτσι ώστε να αναφερθούμε στα άρθρα της οδηγίας και το άρθρο 3 της συνθήκης όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται στο επίκεντρο της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας των πολιτών. Χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας που αποτελεί τον τρίτο πυλώνα ύψης της σημασίας και δεν μπορούμε παρά να εκφραστούμε ελεύθερα και να εκπληρώσουμε το ρόλο μας. Αυτό είναι ένα από τα σημεία τα οποία συμμεριζόμαστε. Γνωρίζουμε ότι η συγγήτρια κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να ανταποκριθούν, όπως είπαν οι συνάδελφοι Χιμένεθ και Ρομέρο, έτσι ώστε να υπάρχει η εποπτεία και η προστασία των θυμάτων. Υπάρχουν χώρες, υπάρχουν συγγνώμη, θύματα τα οποία την χάνουν προστασία στη χώρα τους, αλλά όταν μετακινηθούν από αυτήν δεν έχουν καμία προστασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσχέρειες, γιατί τότε θα γίνουμε και πιο αξιόπιστοι έναντι της κοινή γνώμης. Καλώς. Ευχαριστούμε την κυρία Κώστα. Η κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ. Επειδή είμαι υπεύθυνη από τους φιλελεύθερους για αυτή την πρωτοβουλία μετά, μετά από, σήμερα μετά από πληθώρα συναντήσεων βλέπουμε ότι τα θέματα που αφορούν τη νομική βάση και τη μέθοδο εφαρμογής δεν έχουν ε, οδηγήσει σε αίσιο πέρας, δεν έχουν αποφασιστεί. Εγώ είχα ζητήσει από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να διασαφηνίσουμε μέχρι πού θέλουμε να κινηθούμε. Σήμερα αφού άκουσα τις εισηγήτριες Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση και θα ήθελα να πω ότι με πολιτική θέληση θα μπορούσαμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Διότι το θέμα δεν τέθηκε σε σωστές βάσεις ε, εξ αρχής. Οι πρόβαλαν 20 τροπολογίες για τους εξής στόχους. Για να βελτιώσουμε τη νομική βάση της οδηγίας σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ε, νομικής μελέτης που διενεργήθηκε για να βρούμε μία άκρη και μία θετική έκβαση Επίσης, να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς συντονισμού που προβλέπονται μεταξύ κρατών μελών για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες μέσω εντολής και να διαχειριστούμε καλύτερα αυτή την πλαισίωση έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του και στον τομέα των γλωσσικών. Γι' αυτό ζητούμε την κατάρτιση μητρών για την αυτοματοποίηση της ε, διαδικασίας επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων ε, αρχών. Επίσης θα πρέπει να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ διοικητικών υπηρεσιών που αναλαμβάνουν την εφαρμογή αυτής της εντολής. Με τις τροπολογίες μας ε, προτείνουμε ένα μηχανισμό συνέχειας και επιτήρησης αυτού του πλαισίου για να έχουμε σωστούς στατιστικούς δείκτες που να πλαισιώνουν αυτό το φαινόμενο. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης έτσι ώστε αυτή η πρωτοβουλία να έχει θετική απήχηση σε όλες τις χώρες και να χρησιμοποιήσουμε και τις εξουσίες της ΥΠΑ της εκπροσώπου σε τρίτες χώρες. Αυτοί είναι οι πέντε στόχοι που πλαισιώνουν τις 20 τροπολογίες του, των φιλελευθέρων και θεωρούμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει καμία βελτίωση, γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τις δύο εισηγήτριες, δηλαδή να γίνει μια βελτίωση και στις σχέσεις μας με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, έτσι ώστε να δώσουμε απτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μπιλμπά. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος και από τις δύο επιτροπές να πάρει το λόγο, τότε θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή, την κυρία Κνούτσεν. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άκουσα με ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις Σημαντικό είναι να προστατευθούν τα θύματα οικιακής βίας. Είναι προτεραιότητα της κοινωνίας μας. Γι' αυτό η Κομισιόν από την αρχή υποστήριξε όλους τους στόχους της οδηγίας, όπως δήλωσε η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ επανειλημμένα. Δεν θα επανέλθω στα διάφορα νομικά προβλήματα που έθεσε η Κομισιόν σε προηγούμενες περιστάσεις ε, ούτε στη γραπτή μας γνώμη από τέλος Απριλίου που δόθηκε στο Κοινοβούλιο και επικεντρώνεται στην πρωτοβουλία και το ευρύτατο πεδίο εφαρμογής της που θεωρούμε ότι είναι ευρύτερο αφού πρέπει με βάση τις ποινικέ ε, διατάξεις του άρθρου 82. Το βασικό σημείο της ε, θέσης μας είναι ότι τα μέτρα υπό αυτή την οδηγία ως έχει αυτή τη στιγμή θα πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια της ποινική δικονομίας ε, μετά από τη διάπραξη αξιόπινης ποινική πράξης άκουσα με χαρά αρκετούς ομιλητές σήμερα να λέγουν ότι ίσως θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στη νομική βάση και είμαστε ευτυχείς θα είμαστε ευτυχείς να συνεχίσουμε τη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα γιατί νομίζουμε ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική προστασία θυμάτων ε, βάσει πολιτικής αστικής δικονομίας. Ε, υπάρχουν και κάποιες, δεν υπάρχει δηλαδή επαρκής νομική βάση. Υπάρχουν ενδιαφέροντα επιχειρήματα που στηρίζουν την άποψη αυτή ε, στα επιχειρήματα που ακούσαμε σήμερα. Νομίζω λοιπόν ότι θα δώσουμε συνέχεια πάνω σε αυτό το θέμα. Είμαστε, μας ενδιαφέρει όπως και εσείς να βρούμε πρακτικό δρόμο να συνεχίσουμε σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας που θα λαμβάνονται στα πλαίσια του αστικού δικαίου. Υπάρχουν διάφορα δικαιϊκά συστήματα στα κράτη-μέλη, πρέπει να το σεβαστούμε. Η συνθήκη προβλέπει διαφορετικές διαδικασίες για θέματα ποινικά και αστικά και αυτό επίσης θα πρέπει να το σεβαστούμε. Έχοντας αυτές τις διαφορές κατά νουν, εξετάσαμε πρακτικούς τρόπους για να λύσουμε το πρόβλημα. Η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ το έθιξε το θέμα αυτό αρκετές φορές ήδη και ε, είπε, δεσμεύτηκε στεναρά να λάβουμε σοβαρά υπόψη τη δυνατότητα να βρούμε τρόπους για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας των θυμάτων συμπεριλαμβάνοντας και θέματα αστικού δικαίου. Αυτές οι ιδέες θα, θα αποτελέσουν μέρος του συνολικού πακέτου για τα θύματα που θα υποβάλλουμε κατά το πρώτο εξάμεινο του 2011, ούτως ώστε γενικότερα να βελτιώσουμε την υποστήριξη, την προστασία και τα δικαιώματα των θυμάτων. Πρόθεσή μας είναι αυτό το πακέτο το 2011 να μπορέσει να περιλάβει και συγκεκριμένα μέτρα που θα διασφαλίζουν την επαρκή προστασία θυμάτων που απολάβουν μέτρα αστικής προστασίας και θέλουν να μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος, που είναι και ο πυρήνας της συζήτησης και το επίκεντρο της συζήτησης εδώ. Τώρα αρχίσαμε να κάνουμε τις προπαρασκευαστικές εργασίες που μπορεί να λύσουν και άλλα προβλήματα που αναφέρατε εδώ και που θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε ένα χωριστό μέσο με χωριστά μέτρα που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αστικού δικαίου. Είναι πολύ νωρίς να πούμε ακόμα ποια θα είναι αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα, αλλά ε, για να δείξουμε τη δέσμευσή μας ε, να προχωρήσει η δουλειά, κάναμε μια συνάντηση με τα κράτη-μέλη στα τέλη Μαΐου για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το είδος των περιπτώσεων διοικητικού και αστικού δικαίου που έχουν εξαιρεθεί από την παρούσα πρόταση. Επίσης, είμαστε τώρα στη διαδικασία να κάνουμε μια μελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα καλύψει τις διάφορες εναλλακτικέ για τα θύματα που ενέχονται σε μέτρα αστικής προστασίας για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα τα χάνουν, καθώς θα περνούν τα σύνορα το πόρισμα της μελέτης θα υποβληθεί κάποια στιγμή το φθινόπωρο. Αργότερα, επίσης, κάνουμε μια μελέτη επιπτώσεων για το πακέτο για τα θύματα του χρόνου. Και εκατοντάδες ε, πραγματικά ειδικοί συμμετείχαν και συμμετέχουν με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις για να μάθουμε τη γνώμη τους για το πώς θα οργανώσουμε ένα μηχανισμό νομικό ή μη για θέματα αστικής προστασίας πολιτικής. Ε, επίσης τον Ιούλιο άρχισε δημόσια ε, διαβούλευση για τα θύματα η οποία θα συνεχιστεί μέχρι το Σεπτέμβριο και θέτει σειρά ερωτημάτων που ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν οι ροές που θα μπορέσουμε με τη σειρά μας να βάλουμε μέσα στο πακέτο για τα θύματα. Έτσι λοιπόν ελπίζω ότι αυτά τα μέτρα καταδεικνύουν την προσπάθειά μας να προχωρήσουμε επί της ουσίας και να μην παγιδευτούμε μόνο σε νομικά θέματα. Θέλουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα που θα συνάδουν με τη συνθήκη και τη νομική βάση της νέας συνθήκης. Αλλά είναι σημαντικό να γίνει αυτό μέσα στο σωστό πλαίσιο, ώστε να μην υπάρχουν νομικές επιπτώσεις. Πιστεύουμε ότι ένα χωριστό μέτρο που μπορεί να εκτιλήσεται χωριστά και παράλληλα, με το ποινικό κομμάτι θα είναι ο αποτελεσματικότερος και καλύτερος, βιωσιμότερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα να ακούσουμε τις απόψεις του βελγικού κράτος. Παρακαλώ, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, που δίνετε τη δυνατότητα να εκφραστώ πάνω σε αυτό το θέμα εκ μέρους της Προεδρίας. Πρώτη φορά παίρνω το λόγο σε αυτήν εδώ την αίθουσα να ευχαριστήσω τα δύο μέλη για τον τρόπο με τον οποίο δουλέψανε για αυτό το θέμα αλλά που αφορά και όλα τα θύματα βίας. Με ενδιαφέρον διάβασα και άκουσα επίσης τη συζήτηση σήμερα και διαπίστωσα οι τροπολογίες, οι τροπολογίες που προτείνουν είναι καινοτόμε. Οδηγούν σε μια ενίσχυση της προστασίας του, των θυμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να σας διασφαλίσω ότι το Συμβούλιο καταλαβαίνει πόσο σημαντικός είναι ο διάλογος με το Κοινοβούλιο για να βελτιωθούν οι προτάσεις στις οδηγίες. Η Προεδρία επίσης σας διασφαλίζει ότι η, προστασία των θυμάτων εγκλήματος και κυρίως αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση αποτελούν την προτεραιότητα της ε, Προεδρίας του Βελγίου στη δι... θέματα δικαιοσύνης. Αποτελεί ε, ένα από τα θέματα λοιπόν προτεραιότητας. Επίσης η Προεδρία γνωρίζει ότι αυτό το σχέδιο οδηγίες είναι ένα δύσκολο θέμα αυτή η πρόταση, το βασικό της στοιχείο είναι το πεδίο εφαρμογής και η νομική βάση. Ε, υπάρχουν δύο τάσεις. Μία μειοψηφούσα, η οποία θέλει πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογή και μια μεγαλύτερη τάση που θέλουν ένα μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογή. Η Προεδρία της Ισπανίας έκανε μεγάλες προσπάθειες για να πετυχθεί μια συμβατική λύση και να βρεθεί μια μέση λύση σε αυτές τις δύο προτάσεις. Η τάση λοιπόν μέχρι τώρα ήταν να ενισχυθούν ε, τα θέματα που αφορούν ε, που έχουν να κάνουν με την ποινική πτυχή του θέματος. Επίσης να πω ότι αυτό το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συζητήσεων, μιας μεγάλης συζητήσεως μάλλον, ανάμεσα στους υπουργού όταν τον Ιούνιο είχαμε το Συμβούλιο και στο τέλος του διαλόγου η Ισπανική Προεδρία θεώρησε ότι υπάρχει αρκετή, ε, αρκετή λόγη, να συνεχίσουμε τον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα αποτελεί σημαντικό ουσιώδες στοιχείο για να μπορέσει κανένα να συζητήσει, κανείς συζητήσει σε επίπεδο Συμβουλίου. Εκ μέρους της Προεδρίας τώρα, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας για να ξεκινήσουμε τη συζητήση και να δουλέψουμε μαζί για την επίτευξη μιας συμφωνίας, ούτως ώστε να δώσουμε στα θύματα ένα πλαίσιο ε, προστασίας το οποίο είναι απλό, ε, χρήσιμο και ε, πρακτικό εφαρμοσισμό. Ευχαριστώ, Πρόεδρος να έχουμε τώρα και σχόλια από τις δύο εισηγήτριες. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Χιμινές. Παρακαλώ. Eh. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους καθώς και τη Βελγική Προεδρία και την Επιτροπή διότι ε, προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα και τις προσπαθίες μας. Θα ήθελα να πω ότι επιβεβαίωσα τις ανησυχίες της πλειοψηφίας. Είναι αυτό που είπα από την αρχή. Διότι ένα από τα βασικά ζητήματα δεν έχει επιληθεί Εμείς είδαμε πώς προέκυψε αυτή η εντολή, την είδαμε να γεννάται και ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή η διαδικασία. Συνήλθαμε πολλές φορές με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Το είπαμε και υπό Ισπανική Προεδρία και τώρα υπό Βελγική. Θα συναντηθούμε στις 16 του μηνός με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν έχουμε έναν συνεχή διάλογο. Θα κάνουμε βήματα προς τα εμπρός για να προσεγγίσουμε οι μεν τους δε. Αλλά δυστυχώς ε, θα πρέπει να υπάρχει κάποια κινητικότητα. Δεν, δεν μπορούμε να είμαστε άτεγκτοι. Γι' αυτό μίλησα για τη νομική βάση. Μπορούμε να μιλήσουμε, να γίνει λόγος για το άρθρο 3, αλλά θα πρέπει να ε, υπάρχουν, να βρούμε λόγους ένωσης και όχι απόκλησης των κρατών μελών. Υπάρχουν κράτη που θέλουν να ε, κατοχυρώσουν τις ελευθερίες τους ή να τις ε, διατηρήσουν. Υπάρχουν χώρες που λόγω νομοθεσίας δεν μπορούν να αποδεκτούν αυτό το πλαίσιο. Πολλές φορές υπάρχει εθνικό θέμα και όχι πολιτικών ε, κομμάτων. Κατά τα άλλα εμπλουτίσαμε το περιεχόμενο. Έχουμε νέες βάσεις δεδομένων. Ο κύριος Γιακολίνο είπε ότι δεν θέλει μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά θα πρέπει να τεθεί μια προθεσμία, γιατί πρέπει να δράσουμε τάχιστα. Η ουσία του ζητήματος είναι η εφαρμογή και η νομική βάση και εδώ θα εργαστούμε άοκνα με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, καθώς και με τους συναδέλφους, γιατί το χρωστάμε στα θύματα. Είναι πολύ καλός αυτός ο στόχος, πολύ εύλογος γιατί θέλουμε να διαπρύνουμε το πλαίσιο, αλλά ε, γνωρίζουμε και αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερα εμπόδια. Κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφευχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε ο λόγος περνάει στην κυρία ε, Ρομέρο για ένα τελευταίο σχόλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να πείσω την Επιτροπή όπως πάντα κάνω σε αυτό το θέμα, προς αυτό το θέμα. Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε αυτή την πρωτοβουλία ως παράλληλα μέτρα ή συνοδευτικά μέτρα στο ποινικό δίκαιο σε χώρες όπου επιτρέπεται κάτι τέτοιο δυναμικέ του αστικού δικαίου. Θα μπορούσα όμως να υποβάλω και μία πρόταση οδηγίας. Θα μπορούσε να προβάλλει η Επιτροπή μία πρόταση οδηγίας και εμείς θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε με τροπολογίες. Αυτό το κάναμε σε άλλα πλαίσια όπου συνέβη ακριβώς το ίδιο. Ε, πρόκειται για μία ψευδοσυζήτηση διότι το θέμα της νομικής ε, βάσης δεν είναι θέμα αρμοδιότητας. Δηλαδή, ποιος ε, προβάλλει την πρωτοβουλία η Επιτροπή ή τα μέλη του Συμβουλίου, διότι αν είναι τα μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούμε να ακυρώσουμε μια πρωτοβουλία τέτοιας εμβέλειας. Αυτό θα ήταν μια βαρβαρότητα. Η Επιτροπή προβάλλει μια πρωτοβουλία αλλά ακόμα και αν δεν ήταν έτσι, εφόσον υπάρχει πρωτοβουλία και είναι επίγοντος χαρακτήρα, σε αυτή την περίπτωση η Επίτροπος θα πρέπει να φανεί γενναιόδορη έτσι ώστε να δεχτεί το ίδιο που ισχύει και στην περίπτωση επιδόσεων. αυτό θα μπορούσε να το έχει κάνει, να το έχει προβάλει. Δηλαδή, είναι εντελώς ακατανόητο και δεν καταλαβαίνουμε γιατί η Επίτροπος δεν το δέχεται αυτό. Η ευρωεντολή αφορά την βία κατά των γυναικών. Και αυτό πλήττει όλα τα θύματα γιατί να μην προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα που είναι επίγον. Γιατί βλέπουμε ότι θα έπρεπε να προβάλλουμε μια ειδική εντολή κατά αυτό των θυμάτων οικιακής βίας κυρίως. Γιατί η Επιτροπή δεν το κατανοεί αυτό και οδηγεί σε μια γενικότερη σύγχυση ως προς τη νομική βάση. Ας αφήσουμε αυτό το θέμα και ας ε, δούμε πώς μπορεί να συνεισφέρει η Επιτροπή. Ακόμα βρισκόμαστε στα, σε λογικά πλαίσια. Στις 29 θα πρέπει να ψηφίσουμε. Και θα πρέπει να επικεντρώσουμε το, θέμα μας όχι στη νομική βάση αλλά στις αρμοδιότητες μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής. Δεν είναι δικό μας θέμα, δεν είναι θέμα Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ρομέρο. Να επενθυμίσω ότι η ενδεικτική ψηφοφορία θα γίνει 29 Σεπτεμβρίου που είναι και η επόμενη συνεδρίασή μας πριν να κλείσουμε τη σημερινή κοινή συνεδρίαση θα ήθελα πάρω αυτή, δράξω αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον, ε, τον κύριο Λόπες Αγγιλάρ που συμπρόεδευσε εδώ από την Επιτροπή ε, Δημοσίων Ελευθεριών τη Γραμματεία, όλες οι συναδέλφες και συναδέλφους πολύ σημαντική συνεργασία σε αυτά τα θέματα που είναι κοινά και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα το ότι είχαμε δηλαδή μια τόσο αγαστή συνεργασία. Σας ευχαριστώ λοιπόν και ε, εν γένει ευχαριστώ για τη σημερινή συνεδρίαση και αυτό και εκ μέρους της ε, γραμματείας. Φυσικά να ευχαριστήσουμε και τους ε, διερμηνείς που μας βοηθούν και αυτοί, αυτή την πλευρά τους. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ και επόμενη συνεδρίαση 29 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ. Thank